So, Μετά τον μαραθώνιο των ψηφοφοριών ε, του πρωινού, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και έχουμε μία ακρόαση, οπότε καλωσορίζω τον δόκτωρα Μάρκ Σπρέγκερ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, Υγείας ε, και ασφάλειας ε, των τροφίμων. Χαιρόμαστε για το ότι είστε εδώ πέρα, γιατί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί σας και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία θα συνταχθεί και μια επιστολή με μια σύσταση. Εγώ χαίρομαι επίσης για το ότι καλωσορίζουμε την ε, καθηγήτρια την κυρία Μινέρβα Μαλιόρη που ήταν και ευρωβουλευτής στο παρελθόν και τον ε, καθηγητή τον κύριο Σέρι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καλώς ήρθατε ξανά στο Κοινοβούλιο. Μετά καλωσορίζω τον καθηγητή Ράπτσικ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Είστε ο νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθηγητή Έκταλ που ήταν ο ενδιάμεσος, ο προσωρινός πρόεδρος πρώτης ε, προκατόχου ε, της κυρίας ε, Σουζάννα Γιάκο, Γιάκομπ που ήταν εδώ στην Επιτροπή. Οπότε καλώς ήρθατε όλοι στην Επιτροπή. Ο κύριος ε, Μάρκα ε, Σπρέγγερ ορίστηκε στις 19 Μαρτίου νέος διευθυντής ε, της υπήρεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη στην Στοχόλμη Δεν είστε άγνωστος. Ήσασταν και εσείς επικεφαλής του διοικητικού αυτού συμβουλίου. Θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο ότι από τη δεξιά πτέρυγα πήγατε στην αριστερή και ταυτόχρονα ήσασταν διευθυντής ε, στην Ολλανδία του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος και ασχοληθήκατε επί σειρά ετών με αυτά τα θέματα. Η Επιτροπή μας λοιπόν ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με τα θέματα υγείας, είναι τομές ευθύνης μας και έχουμε μέλη που παρακολουθούν πάρα πολύ στενά όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τα της υγείας και βέβαια παρακολουθούμε και το έργο του κέντρου σας όπως και η Κομισιόν άλλωστε στον τομέα της πολιτικής ε, υγείας. Βεβαίω έχετε εκεί ένα διεθνές ε, περιβάλλον ε, ανθρώπους από διάφορες χώρες, πρέπει να συνεργαστούν, πρέπει να τους δώσετε κίνητρο. Στη Στοκχόλμη βεβαίως η Στοχόλμη είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα πόλη, δεν ξέρω αν καταφέρετε να βρείτε ανθρώπους για να έρθουν ε, εκεί πέρα. Δεν θα, δεν θα ρωτήσω εγώ τώρα τα πάντα για την κάθε αρρώστια ξεχωριστά, ούτε για τη φυματίωση, ούτε για τίποτα άλλο. Σας δίνω τον λόγο λοιπόν να κάνετε την παρουσίασή σας. Members of this committee, it's really great honor. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είναι τιμή μου να μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ ενώπιον σας σήμερα. Ξέρω ότι η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη από Ιδρύσεώς της, η Σουζάννα Γιάκαμπ, εκτιμούσε ιδιαίτερα την υποστήριξη της Επιτροπής σας όταν ήταν στα Σπάργανα ο οργανισμός. Ελπίζω να συνεχίσετε λοιπόν να αγαπάτε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη τώρα που μπαίνει στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος της ζωής μας και ε, είναι όμως και ταυτόχρονα και μια πολύ ζωντανή και μια περίοδος που σε ε, ανταμείβει. Έχω εμπειρία γιατί έχω τέσσερα παιδιά στην εφηβεία. Προσβλέπω λοιπόν ε, στις συμβουλές σας και θα απαντήσω και τις ερωτήσεις σας εντός ολίγου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω λίγα πράγματα για μένα και το τι ακριβώς σχεδιάζω για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη. Ε, σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ και εκεί μου έμαθαν την έννοια του υγεία για όλους. Αυτό ε, μου έδωσε και την αίσθηση που έχω για τη δημόσια υγεία έκτοτε. Ε, στη συνέχεια ειδικεύτηκα ως μικροδιολόγος και έκανα και ένα διδακτορικό στην επιδημιολογία της γρήπης. Ναι, η γρήπη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η εμπλοκή μου στην πολιτική υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε περίπου πριν από 20 χρόνια, όταν ήμουν επικεφαλής ε, του Επιδιομολογικού Κέντρου Λιμωδών Νόσων ε, στο ε, Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας ε, της Ολλανδίας και συμμετείχα και σε μια ομάδα ενθουσιωδών ανθρώπων που με υποστήριξη της ευρωπαϊκή επιτροπή, άρχισαν να δημιουργούν δίκτυα εμπειρογνωμόνων που ε, διασύνδεαν τη δημόσια υγεία ανά την Ευρώπη. Προσπαθούμε να έχουμε, προσπαθούσαμε να έχουμε καλά στοιχεία συγκρίσιμα για ε, μολυσματικές ασθένειες όπως η φυματίωση, το AIDS, η πατήτιδα, η οποία είναι ακόμα πολύ σημαντική και την νόσο των λεγιονάριων. Αυτή η δουλειά που έγινε στη δεκαετία του 90 μας βοήθησε να αποδείξουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά των μολυσματικών ασθενειών και ορισμένοι από εμά ε, σκεφτόμασταν ήδη ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης τότε. Ω διοικητικό τέλεχο άρχισα να εργάζομαι περίπου πριν από 7 χρόνια, όταν έγινε Γενικό Διευθυντή ε, του Ολλανδικού Εθνικού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Μιλάμε για ένα Ινστιτούτο το οποίο αριθμεί περίπου 1.500 μέλη προσωπικού και έχει και ένα ετήσιο προπολογισμό τη τάξη των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από 7 χρόνια στο τιμόνι του οργανισμού αυτού, μπορώ να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά την δημόσια υγεία και ξέρω πώ μπορώ να ηγούμε ενό μεγάλου πολύπλοκου οργανισμού σε ένα περίπλοκο ε, πολιτικό περιβάλλον. Γνωρίζω λίγο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Πρόληψη, κυρίως πόσο υψηλές και πόσο ποικιλόμορφες είναι οι προσδοκίες ε, για τον οργανισμό αυτό από τους ενδιαφερομένους. Μέχρι πριν από δύο χρόνια ε, προέδρευα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, δηλαδή ήμουν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ξεκίνησε το κέντρο και ε, καθορίστηκαν οι στρατηγικές του κατευθύνσεις. Όσον αφορά στις προτεραιότητές μου, ε, καταρχάς με τιμά το γεγονός ότι το περασμένο μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου με εξέλεξε να είμαι επικεφαλής του Κέντρου και τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντική περίοδος για το Κέντρο. Κληροδοτώ ένα κέντρο με ε, εξαιρετικό προσωπικό, ε, με μεγάλη διάθεση για εργασία και εξαιρετική ε, φήμη. Θέλω να παγιωθούν τα επιτεύγματά του και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω. Δεν σκοπεύω να κάνω άμεσες αλλαγές ε, στις επιστημονικές προτεραιότητες του κέντρου, οι οποίες ε, επισημάνθηκαν από τη Σουζάννα Γιάκαμπ και σας τις παρουσίασε και το Σεπτέμβριο. Οι βασικές προκλήσεις λοιπόν για τη δημόσια υγεία του κέντρου εστιάζουν και θα συνεχίσουν να περιλαμβάνουν την αντιμικροβιακή αντοχή, το AIDS, την φυματίωση, τις αναδυόμενες νόσους την αλλαγή του κλίματος και φυσικά τη γρήπη. Τώρα, βλέποντας λίγο προς το μέλλον, σκοπεύω να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία εγκάρσια θέματα, τρεις προκλήσεις από διοικητικής πλευράς. Καταρχάς να διασφαλίσω ότι η αριστεία των γνωμοδοτήσεων του, που δίνει το ECDC θα εξακολουθήσει να υφίσταται και δεύτερον να ενισχύσω περαιτέρω τις ε, βασικές εταιρικέ μας σχέσεις. Τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχει καλά αποτελέσματα ο οργανισμός ε, ως ευρωπαϊκός αποκεντρωμένος οργανισμός. Καταρχάς λοιπόν η επιστημονική αριστεία. Αυτό βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου μου. Θέλω ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πρόληψη να είναι ο πρώτος οργανισμός που σας έρχεται κατά νου όταν θέλετε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τις μολυβηματικές ασθένειες. Θέλω να είστε 100% βέβαιοι ότι οι γνωμοδοτήσεις που λαμβάνετε είναι έγκυρες, ανεξάρτητες και βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Όταν θα ε, εκπονούνται οι γνωμοδοτήσεις μας θα κάνουμε ευρεία διαβούλευση και θα μιλάμε με ένα μεγάλο φάσμα εξωτερικών εμπειρογνωμών. Ωστόσο, θα σας λέμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονε και κατά πόσον υπάρχουν και αντικρουέμενα συμφέροντα η τελική απόφαση για το τι γνωμοδοτήσεις ε, δίνει το ECDC ε, θα είναι δική μου αρμοδιότητα ως διευθυντής ε, του κέντρου. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις, αυτές είναι ένα απόσπαστο τμήμα του ECDC γιατί βασιζόμαστε στους πόρους και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Θέλουμε να έχουμε ισχυρά αποδοτικά δίκτυα τα οποία θα τα διατηρούμε με τα κράτη-μέλη. Και κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, θέλουμε να έχουμε εταιρικέ σχέσει με του ενδιαφερομένου στι χώρε γείτονε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έχουμε, ακόμα, έχουμε ήδη εξαιρετική συνεργασία με τον ΠΟΗ και αυτό φυσικά θα πρέπει να παραμείνει και θα πρέπει να ενισχυθεί θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με άλλους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των ε, Τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Οργανισμό της Κοπενχάγης. Ε, βέβαια, οι πιο σημαντικές εταιρικέ μας σχέσεις είναι με τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, το Συμβούλιο και φυσικά εσάς περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τις ε, προτεραιότητες ε, που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της πρόληψης, διότι το ECDC θα πρέπει να υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν σήμερα να είναι η αρχή ενός παραγωγικού διαλόγου και να δημιουργηθεί μια ε, σταθερή εταιρική σχέση μεταξύ μας. Τώρα, όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα. Η τρίτη και τελική προτεραιότητα είναι να διασφαλίσω ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Πρόληψη είναι ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο εταίρο για του ενδιαφερομένου μα. Θέλω να μπορώ να προσλαμβάνω και να ε, προσωπικό υψηλού επίπεδου το οποίο θα παραμένει στον οργανισμό και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός θα δίνει εξαιρετικές ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Θέλω να μπορώ να επενδύω στο προσωπικό μου και να τους προσφέρω καλές συνθήκες εργασίας που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να τους προσφέρουμε καλές συνθήκες διαβίωσης στη Σουηδία. Το να υπάρχει μια καλή συμφωνία ως προς την έδρα με την χώρα που μας φιλοξενεί είναι συνεπώς ε, προτεραιότητα για μένα και μάλιστα από την αρχή. Πέραν αυτού, ξέρω ότι ζούμε σε καλεμπούς καιρούς, ο, οι προπολογισμοί για την υγεία είναι υποπίεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό ακριβώς και το ECDC θα πρέπει κάθε ευρώ που δαπανά να, το δαπανά σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει ε, κατάλληλη λοιπόν σχέση κόστους ωφελίας και να υπάρχει και αριστεία. Το αναγνωρίζω αυτό και φυσικά είμαι υπόλογος και προς όλους εσάς για το θέμα αυτό. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, σκοπεύω να συνεργαστώ με τους ενδιαφερομένους του ECDC και και ιδιαίτερος της Επιτροπής σας και θέλω να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να συνεργαστούμε ώστε το όνειρο της υγείας για όλους να υλοποιηθεί βαθμιδών από κοινού και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις γείτονες χώρες, διότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό ακριβώς ε, και έκανα αίτηση για να κάνω αυτή τη δουλειά και γι' αυτό ακριβώς βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Σπρέγγερ, για την ε, εισαγωγή σας σε αυτή την ε, μικρή ακρόαση. Ακούσαμε τη δική σας παρουσίαση και οι συνάδελφοι θα κάνουν τις ερωτήσεις. Η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη είναι το άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή και η ομάδα την οποία εκπροσωπεί θα ξεκινήσει τώρα με τον Πέτερ Λίζε. Τρία λεπτά έχουμε, ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε δόκτωρ Σπρέγκερ για την ε, παρέμβασή σας. Και θα ήθελα πριν να κάνω την ερώτησή μου να υπενθυμίσω σε όλους ε, την συνεισφορά του John Bowis, που ήταν ε, αυτός που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων με μεγάλη ανάληψη δέσμευσης και αφοσίωση ε, προχώρησε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η δική σας εικόνα για το ECDC, ποιο είναι το όραμά σας για το περιβάλλον και την υγεία μα ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά και η σύνδεση μεταξύ αυτών των θεμάτων. Στην ακρόαση το Σεπτέμβριο η Σουζάνα Γιάκοψ είχε αναφέρει εν συντομία ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων θα εργαστεί και σε θέματα κλίματος και υγείας, αλλά συγκεκριμένα τι προβλέπετε, τι σενάρια υπάρχουν, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για την πολιτική που θα ακολουθήσετε. Και δεύτερον, μια έρευνα της British Medical Journal τους τελευταίους μήνες ε, μεταξύ των αναγνωστών του British Medical Journal, δηλαδή κάποιοι που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ιατρικά θέματα, ε, ρωτούσε για θέματα αντιμετώπισης νόσων και ε, φάνηκε ότι το κύριο μέλημα είναι το καθαρό νερό, ούτε αντιβιωτικά ούτε τίποτα άλλο. Μήπως θα ήταν καλύτερο μέσω πρόληψης των λιμωδών νόσων λοιπόν το να αποφεύγουμε νόσους που μεταδίδονται μέσω του νερού. Ευχαριστούμε τον Πετελίζε. Ε, είπα προηγουμένως ότι είμαστε σε ακρόαση και πρέπει να πω ότι έχουμε σαν ένα παιχνίδι πινκ-πονγκ, όχι τρία λεπτά, δηλαδή ένα-δύο λεπτά ο καθένας για να μπορούμε να έχουμε την απάντηση κατευθείαν από τον ομιλητή. Σας δίνουμε το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Λίζα. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε και στην αλλαγή του κλίματος και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω δύο λόγια από αυτού. το θέμα της κλιματικής αλλαγής ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερος και αυτή τη στιγμή η συζήτηση ε, γίνεται μεταξύ εμπειρογνώμων σχετικά με το περιβάλλον. Όπως το βλέπω εγώ, η συζήτηση δεν είναι στα χέρια των Υπουργών Υγείας και θα ήθελα η κλιματική αλλαγή περισσότερο να μπει στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Υγείας. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Γνωρίζουμε όμως με τα βεβαιότητες ότι οι λοιμώδεις νόσοι θα επηρεαστούν από την αλλαγή του κλίματος. Αναφέρατε και το νερό. Και το νερό θα επηρεαστεί και κατά ποικίλου τρόπους θα μπορούσε να επηρεαστεί το νερό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές αβεβαιότητες. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος που το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συγκεντρώνει πολλές πληροφορίες. Συνδυάζει πληροφορίες από πολλές πηγές και περιβαλλοντικές πηγές και πηγές από τον τομέα της υγείας. Ξεκίνησαν τώρα το πρόγραμμα ε3 ε, ε, ε, που, που συνδυάζει όλα αυτά τα δεδομένα και χαίρομαι ιδιαίτερος διότι ότι ένα βασικό άρθρο στο Lancet ε, αφορά τις δραστηριότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης. Διεξάγει λοιπόν πολλές μελέτες στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης για να δούμε πόσο ευάλωτοι είμαστε στην κλιματική αλλαγή. Έχουμε το πρόγραμμα ε3 που συνδυάζει δεδομένα από πολλές πηγές και επίσης δίδουμε στα κράτη-μέλη ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν θέματα στα οποία είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις της κλίμακας, ε, όπως είναι ένα, ένας ιός στη Δυτική Ευρώπη που προκαλείται από κουνούπια που μπορούν να επιβιώσουν στο νερό και ο πυρετός Ντέγκε είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και υπάρχουν και οι νόσοι που μεταφέρονται από τσιμπούρια και ε, αυξάνονται σιγά σιγά και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στις περιβαλλοντικές πτυχές της αλλαγής του κλίματος αλλά θα πρέπει να απασχολήσει και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας. Στο μέλλον λοιπόν προσβλέπω σε συζητήσεις μαζί σας και ελπίζω να το θέσετε σε προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η Dagmar roth Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα πως ε, διαβάζετε και καταλαβαίνετε γερμανικά κύριε Σπρέγκερ, οπότε θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις στα γερμανικά. Πρώτα απ' όλα κάποιες που αφορούν εσάς και μετά την υπηρεσία. Χαρήκατε για το ότι σας όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος αν δεν θα συζητήσω την ε, διαδικασία. Ξέρετε πως είχε ασκηθεί κριτική από την Κομισιόν για την διαφάνεια του ΔΣ. Θεωρείτε πως, πως θα έχετε τη στήριξη του ΔΣ και πως θα είναι ο ρόλος σας εκεί πέρα. Είπατε πως ήρθατε εδώ πέρα να ακούσετε συμβουλές. όταν μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν το στυλ ε, της διοίκησής σας δεν τους ήρθε αυτό ε, έτσι ως ε, το πρώτο χαρακτηριστικό σας. Θεωρείτε λοιπόν ότι ασκείται η ηγεσία συμπεριλαμβάνοντας τους άλλους και μπορεί να, μπορείτε να τους κινητοποιήσετε ή είστε κάπως πιο έτσι αυταρχικός και ιδιαίτερος στο στυλ σας. Επίσης, όσον αφορά τα συγκρόμενα συμφέροντα. Είπατε πως είστε διευθυντής ενός μεγάλου Ινστιτούτου και είπατε πως είναι μεγάλο. Θεωρείτε πως είναι σωστό ο πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου να συναποφασίζει ε, το δικό του Ινστιτούτο να λαμβάνει ένα έργο που κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Γνωρίζω πως τα Εθνικά Ινστιτούτα λαμβάνουν χρήματα, αλλά θεωρείτε πως ε, θα είναι άμεμπτο ας πούμε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση δηλαδή όταν ο πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου στέλνει ξέρω εγώ συμβόλαια μισού εκατομμυρίου ευρώ επί σειρά ετών στο Ινστιτούτο Εγώ δεν το βρίσκω. Εντάξει και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για τα αντικρώμενα αυτά συμφέροντα και το τι θα κάνετε στο μέλλον εάν ε, προκύψουν αναλογές καταστάσεις. Κατόπιν θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για τον ρόλο του ECDC. Προέρχεστε από μια μεγάλη κρατική αρχή και είστε περήφανος ε, και δικαίως, αλλά έχετε καταλάβει ότι πρόκειται περί Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας, το, το ECDC. Έχετε εδώ πέρα αφεντικά χρηματοδοτήστε 100% από τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οπότε προβλέπετε ότι θα ακολουθείτε αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν και η προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τελευταία μου λέξη, κύριε Πρόεδρε, τι θεωρείτε ε, πως έχει κάνει μέχρι στιγμής όσον αφορά το κέντρο σας, όσον αφορά την προσθέμενη αξία και στην πράξη και στην ε, νομοθεσία. Και θα επανέλθω κύριε Πρόεδρε γιατί έχω πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Σπρέγκερ. Εμφανίζεται ακόμη δύο φορές ε, στον κατάλογο των ομιλητών, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, πατήστε το κουμπάκι και ανοίγει το μικρόφωνο. Um, Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι δύσκολο να κρίνω εγώ ο ίδιος ε, το δικό μου ύφος στο Ινστιτούτο μου, στο RIVM. Μπορώ να σας πω ότι επικρατεί πολύ καλή ατμόσφαιρα και έχω απολύτως τη δυνατότητα να ακούω τις συμβουλές ε, των διευθυντών μου. Ένα είναι ο κ. Σκουτίγιο που μιλά πολύ ανοιχτά και έχω μάθει πως... Επίσης, ε, με χαρά άκουσα τις απόψεις που μου ε, έχει εκφράσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλές φορές ήταν διστάμενες απόψεις και πολλά τα οποία αναμένονταν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο πρόληψη υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες και δεν είναι εύκολο να καλύψει κανεί ε, τι ε, προσδοκίε όλων γιατί ε, οι μεγαλύτερες χώρες μερικέ φορέ έχουν μεγαλύτερε προσδοκίε, οι μικρότερε χώρε είναι πιο ικανοποιημένε από τι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να χειρίζεται κανεί τι αντι... προσδοκίε προσδοκίες όλων. Όσον αφορά τα συγκρουόμενα συμφέροντα, στο μέλλον θα ήθελα να βασιστούμε στη λειτουργία ευρωπαϊκών Ινστιτούτων που είναι πάρα πολύ σημαντικά στον τομέα της δημόσιας υγείας Πολλοί έχουν ζητήσει να έχει δικά του εργαστήρια το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη. Εγώ είμαι υπέρ του να μην έχουμε δικά μα εργαστήρια. Ε, δαπανούμε πολλά χρήματα φορολογουμένων για να δημιουργούνται εργαστήρια, πολύ ωραία εργαστήρια, σε άλλε χώρε. Ήμουν στο Βερολίνο και στο Βερολίνο κατασκευάζεται ένα καινούριο εργαστήριο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Α μην δημιουργηθεί λοιπόν άλλο τέτοιο εργαστήριο και υπάρχει επικάλυψη και στη Στοκχόλμη. Έχουν γίνει ερωτήσεις και για κάποια προγράμματα. Εγώ δεν ήμουν υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ανάθεση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και οι συμβάσεις δόθηκαν στο Ινστιτούτο μου ή σε άλλο Ινστιτούτα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του εκτελεστικού διευθυντού και όχι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομολογώ ότι έχω μεγάλα προβλήματα στην Ολλανδία με το θέμα αυτό διότι σε πολλά εθνικά Ινστιτούτα Δημόσιας Υγείας κοστίζει πολλά χρήματα, πολύ περισσότερα κοστίζει να κάνουν τη δουλειά που τους ανατίθεται σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνουν. Ελπίζω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που λαμβάνουν χρήματα των φορολογουμένων θα συνεργαστούν στην Ευρώπη για την καταπολέμηση των λιμωδών νόσων. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, Αυτό φάνηκε και από την εξωτερική αξιολόγηση. Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο πρόληψη θα δώσει δεδομένα για ανάληψη δράσης και η ανάληψη δράσης στη συνέχεια είναι βέβαια αρμοδιότητα των κρατών μελών, ε, μέρη του Συμβουλίου, της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη ε, δίνει συμβουλές, στοιχεία και πρακτική υποστήριξη στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι πριν από δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης εξέδωσε την πρώτη έκθεση, επιδημιολογική έκθεση για λοιμώδεις νόσους και μας δίνει μια εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε τώρα ποια είναι τα ισχυρά σημεία και ποιες είναι οι αδυναμίες της Ευρώπης και αυτό, αυτή η έκθεση ήταν πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να καταστρώσουμε την πολιτική μας στη συνέχεια. Επίσης, πριν από 10 χρόνια υπήρχαν πολλά διαφορετικά δίκτυα. Ένα δίκτυο για την Legionella, ε, ένα για το HIV κλπ. Και μεταφέρθηκαν υπό την αγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη, και έτσι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά λιγότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν όταν δεν καλύπτονταν από τη γενικότερη αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη. Τα επιτεύγματα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη είναι εντυπωσιακά και νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι έχει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι προφανέ και από την εξωτερική αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Μαρίνα Παρβανόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντώνια Παρμανόβα, η Μαρίνα Γιανακιουδάκης είναι εκεί. Μας μπερδεύουν συνεχώς. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας ε, και για τις απαντήσεις που έχετε ήδη δώσει. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, η ανεξαρτησία της εμπρογνωμοσύνης. Επανειλημμένως ε, για διάφορες ε, νόσους ε, χρησιμοποιούμε τις εκθέσεις και την εμπειρογνωμοσύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι εξωτερική ανάθεση σε διάφορους μη κυβερνητικού οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιστημονικούς φορείς κλπ. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή όπως ακριβώς το κέντρο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε για την πρόληψη. Η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με αυτό. Πριν από κάποιες εβδομάδες εγκρίναμε την ε, έκθεση για τη δράση κατά του καρκίνου, η οποία έχει και ένα εδάφιο που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόμων ε, για τις ε, μη μεταδιδόμενες ασθένειες και να τις συμπεριλάβει και αυτό στην εντολή του. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Τα τελευταία δέκα χρόνια συζητάμε για μεταδιδόμενες και μη μεταδιδόμενες ασθένειε και επίδραση που έχουν στη δημόσια υγεία. μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ανισότητε στην υγεία. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση την οποία θα εξετάσουμε, την οποία θα παρουσιάσει η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πολλές φορές έχουμε θέματα που αφορούν στον καρκίνο, στο διαβήτη, αλλά δεν υπάρχει μια συστημική προσέγγιση για όλες τις νόσους. Θα ήθελα να ξέρω την αποψή σα από αυτού και η τρίτη με ερώτηση είναι μάλλον πρόταση. να έχουμε τις εκθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης για τους εσωτερικούς ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να δούμε τι λένε για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη, ώστε να γνωρίζουμε λίγο και τι έχουν να μας πούν αυτοί. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε, έχετε τον ίδιο χρόνο όσο και ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Αξιοπιστία, διαφάνεια, ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. και έχουμε και κάποιες ad hoc επιτροπές για κάποια θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται ο κώδικας διοντολογίας σε όλα τα μέλη αυτών των ad hoc επιτροπών και να βλέπουμε κατά πόσον υπάρχουν και αντικρουέμενα συμφέροντα. Εάν υπάρχουν, τότε φροντίζουμε να αποφασίσουμε κατά πόσον μπορούν να συμμετέχουν ή όχι στην ε, κάθε επιτροπή. Υπάρχει και ένα συμβουλευτικό φόρουμ και στο φόρουμ αυτό υπάρχουν πάρα πολλά μέλη, εμπειρογνώμονες ε, σε θέματα δημόσιας υγείας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΠΟΗ και από διεθνείς οργανώσεις ε, για την υγεία και θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Η τελική απόφαση ούτως ή άλλως επαφίεται στον Γενικό Διευθυντή για τις γνωμοδοτήσεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαφάνεια και θα ήθελα στην ε, ιστοσελίδα να υπάρχει και η δήλωση ε, οικονομικών συμφερόντων γιατί ακριβώς θέλουμε να έχουμε την ε, διαφάνεια που σας ανέφερα. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είμαι διευθυντής ε, του Εθνικού Ινστιτούτου και ξέρω ότι από θέματα υγείας οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες είναι πολύ σημαντικές. Ε, η παχυσαρκία, ο καρκίνος ε, και η φυσική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη γύρανση του πληθυσμού κιόλας. Ε, δεν έχει συζητηθεί ακόμα αυτό το θέμα και δεν, δεν έχουμε δει αν πρέπει να συμπεριληφθεί στην εντολή. Το συζητήσαμε πριν από δύο-τρία χρόνια και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε τουλάχιστον προ το παρόν στι μεταδιδόμενε ασθένειε. Και αυτό με χαροποιεί. Σα είπα στην αρχή τη παρουσίασή μου ότι είμαστε στην εφηβεία και νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να επικεντρωθούμε στι μεταδιδόμενε ασθένειε και από εκεί και πέρα στο μέλλον και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί η εντολή μας. Αλλά κατ' εμέ για λόγους αξιοπιστίας, εάν επεκτείνουμε την ε, εντολή μας, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε πάντα αξιόπιστοι και θα πρέπει να έχουμε και κατάλληλα μέσα και πόρους, ώστε να έχουμε αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν, χρειαζόμαστε και τους εμπειρογνώμονες, αλλά προβλέπω στο μέλλον σε συζήτηση αυτού του θέματος. Όσον αφορά τώρα την πρότασή σας, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα να σας δοθούν τα σχετικά έγγραφα. Και τώρα, όχι η Αντωνία, αλλά Μαρίνα, για να κουδάκι, που είστε και το άτομο που είναι αρμόδιο για την επαφή μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που είπατε σωστά και το όνομά μου. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, ε, Δ. Σπρέγγερ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, διότι υπάρχει αύξηση παγκοσμίω ε, στον αριθμό των γυναικών ε, που ε, υποφέρουν από HIV. Ε, πάνω από ένα εκατομμύριο στον Ηνωμένο Βασίλειο, οποίο είναι το 30% ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο από το 1993 μέχρι το 2008 η αύξηση για τις γυναίκες ήταν διπλάσια. Είναι σημαντικό λοιπόν το πρόβλημα της αύξησης. Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στο AIDS ε, έκανε ένα σεμινάριο που εστιάστηκε στο, στον του AIDS και στους άνδρες. Στο μέλλον έχετε προβλέψει σεμινάρια ή ε, συνέδρια που θα ασχοληθούν με το θέμα του πώς επηρεάζονται οι γυναίκες και πώς θα μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε το πληθυσμό για αυτό το πρόβλημα. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Έχω όμως πάλι ένα λεπτό για να απαντήσω, παρότι ήταν σύντομη ερώτηση. Ωραία, πολύ καλά, ευχαριστώ. Κυρία Γιανακουδάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν διότι προεδρεύσατε στο σεμινάριο πέρυσι για το HIV. Και ανησυχώ ακόμη περισσότερο, διότι μόνο 30% των ατόμων που έχουν ε, μολυνθεί γνωρίζουν ότι ε, είναι φορείς και η πλειοψηφία όπως καταλαβαίνετε δεν το γνωρίζει. Υπάρχει αύξηση σε νέα κρούσματα. Δεν γνωρίζω αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αύξηση μεγαλύτερη για τις γυναίκες. Ε, ξέρω ότι ε, ε, υπάρχει αύξηση σε πολλά νομίσματα για τους χρήστες ναρκωτικών. Ξέρω λόγω των ενδοφλέβιων, της ενδοφλέβιας χορήγησης υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος για την αύξηση αυτή μεταξύ των γυναικών. Θα το ελέγξουμε πάντως. Χαίρομαι που υπάρχει η δήλωση του Δουβλίνου και έχει συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, στη δήλωση αυτή και παρακολουθούν την εξέλιξη του θέματος. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θέλει να ξεκινήσει μια μελέτη βιωσιμότητας ε, για την ε, παρακολούθηση των συμπεριφορών και αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει όσον αφορά την εξάπλωση του HIV. θέλουμε να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα ε, να ελέγχονται και να ε, υποβάλλονται σε θεραπεία για τον HIV και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, προσεχείς περιόδους. Η κυρία Κώστετς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, μα είπατε ότι είστε ειδικό σε θέματα γρήπη. Πριν από λίγου μήνε μιλούσαμε πολύ για τον ιό H1N1 και τώρα πια δεν το συζητάμε. Ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει για τον επόμενο χειμώνα. Τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, μέτρα που δεν έχουν ληφθεί, μέτρα που δεν ελήφθησαν σωστά τους τελευταίους μήνες για να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε προληπτικά τη γρήπη Ακόμη αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ευρώπη οδήγησαν πολλές φορές σε αμφιβολίες όσον αφορά τα εμβόλια και το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, δεδομένου ότι μία από τις βασικές ε, μεθόδους πρόληψης είναι ο εμβολιασμός. Πείτε μας λοιπόν πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα για το μέλλον και πώς μπορούμε να πληροφορούμε καλύτερα τους πολίτες της Ευρώπης για αυτή τη μέθοδο πρόληψης, τον εμβολιασμό δηλαδή, και πείτε μας ε, πώς βλέπετε το μέλλον σχετικά με τη γρήπη. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για την απάντηση. Δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσει κανείς σε αυτήν την ερώτηση. Καταρχήν, η γρήπη αυτή ήταν μια επιδημία χωρίς προηγούμενο. Δεν είχε δηλαδή συμβεί στο παρελθόν. Και τα διδάγματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε από την κατάσταση αυτή είναι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για απρόβλεπτες επίγουσες καταστάσεις. Ήμασταν προετοιμασμένοι για τη γρήπη. Τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν έτοιμα να καταστρώσουν τα προγράμματα για την πανδημία και αυτό αποτελεί μια επιτυχία αλλά είναι πολύ δύσκολο ε, να ε, μεταφέρουμε ε, στο κοινό τα θέματα που έχουν σχέση με κίνδυνο, γιατί υπήρξε μια μεγάλη φοβία σε σχέση με την γρήπη και στην Ολλανδία είχαμε μια τέτοια φοβία που επικράτησε για την γρήπη. Ανησύχησαν πολύ οι πολίτες και πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να έχουμε ισορροπημένη πολιτική επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό δίδαγμα που μπορούμε να πάρουμε. Και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για να ε, έχουμε σωστές ε, συμβουλές πρέπει να είναι πιο διαφανής η διαδικασία. Είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τους γονείς αν μιλάμε για τα εμβόλια στα παιδιά ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Σχετικά με την γρήπη κάναμε κάποιες μελέτες. Τα προκατακτικά αποτελέσματα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα 70% και αυτό σημαίνει ότι το εμβόλιο ήταν σε θέση στο 70% των ε, περιπτώσεων ε, να εμποδίσει ε, αλλαγή του ιού ε, και ε, νόσο των πολιτών, κάτι το οποίο δεν ήταν πάντοτε εύκολο να είναι αντικείμενο της πολιτικής επικοινωνίας μας. Κάναμε πολλές μελέτες και Τώρα είναι σαφές ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητος, διότι στην Ολλανδία δώσαμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του νέου εμβολίου για τη γρήπη και ήταν απολύτως ασφαλές. Δεν υπήρχαν παρενέργειες και δεν αναφέρθηκαν σχεδόν καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες. Η κυρία Ντάκμα Ροτ Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπα πριν. Δεν με πείσατε κύριε Σπρέγγερ, αλλά ίσως δεν ξέρω αν το περιμένατε. Δεν με πείσατε με το να λέτε πως τα εμβάσματα σε εθνικά Ινστιτούτα είναι βάρος αντί για όφελος. Άμα είναι έτσι, ας τα αφήσουμε το ECDC και να πάνε τα λεφτά κατευθείαν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε για κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό ότι όπως και κάθε άλλη υπηρεσία θα βάλετε στην ιστοσελίδα σας τα οικονομικά συμφέροντα των μελών σας και πως τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ που ταυτόχρονα εργάζονται σε εθνική υπηρεσία και στο πλαίσιο του ΔΟΥΣΟΥ έχουν πρόσβαση σε έργα ή συμμετέχουν σε έργα ή αποφασίζουν για έργα που έχουν βεβαίως ε, χρηματικό αποτέλεσμα και αυτά θα δώσουν τα οικονομικά τους ε, συμφέροντα. Εσείς είπατε για το δικό σας το, το Ινστιτούτο. Και το, πόσα, το ότι λαμβάνει κάθε χρόνο ε, μισό εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχουν ε, εργαστήρια, εντάξει. Αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα δεν ξέρω αν έχει νόημα. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν είναι και τόσο διαφανές αυτό το οποίο κάνετε εσεί στο Χόλμ. Εγώ θα ήθελα διαφάνεια. Επίσης για τα επιτεύγματα. Είπατε πώς τα επιτεύγματα σας είναι εντυπωσιακά. Η κυρία Τζέικομπ ε, από μένα άκουγε χρόνια πως δεν με εντυπωσίαζε τόσο πολύ. Και αναμένω ακόμα να με πείσει κάποιος ε, τι είναι ακριβώς αυτά τα επιτεύγματα. Δηλαδή μπορεί τα δεδομένα τα οποία μαζεύεται να είναι σημαντικά για κάποιες χώρες όπως ε, είναι π.χ. τα στοιχεία του ΠΟΗ αλλά π.χ. για την ε, γρήπη των χείρων. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς επηρεάζεται και ασκείται γρηγορότερα η πολιτική μας και δεν με έχετε πείσει ακόμα το ότι αξίζει το κέντρο σας εντός ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης ε, έτσι ώστε τα επόμενα, αν έχετε ένα σχέδιο δράσης ε, και νομοθετικό, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια πραγματικά να αυξήσετε την, την προσθέμενη αξία σας. Μάλιστα, η προσθέμενη αξία του ECDC για την Ευρώπη. Λοιπόν, όσον αφορά, όπως είπατε, την σύγκριση συμφερόντων. Υπάρχει σχετική δήλωση, έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα για όλα τα μέλη του ΔΣ, εμού συμπεριλαμβανομένου και έχουμε δημοσιεύσει και ένα φύλλο με όλα τα χρήματα τα οποία λαμβάνουμε από ε, οπουδήποτε ε, είτε από το ECDC είτε από οπουδήποτε άλλο. Οπότε είναι σαφές ε, και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αδιαφάνειας όσον αφορά τα χρήματα που έλαβε το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της ε, Ολλανδίας. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, μιλώντας και για την γρήπη, νομίζω επιδείξαμε πως ε, προσπάθησα να το δω από μια εθνική σκοπιά ενός κράτους μέλους. Για μας ήταν εξαιρετικά σημαντικό κάθε μέρα να έχουμε τις καινούριες πληροφορίες για την επιδημία. Και αυτές τις πληροφορίες τις έδινε το κέντρο μας. Και έκανε και την αξιολόγηση κινδύνου. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό σε εθνικό επίπεδο. Και βεβαίως σε εθνικό επίπεδο ο Υπουργός Υγείας εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο ε, για τον δε τον δε των ε, θυλωμάτων. Θυλωμάτων. Εμείς ε, δώσαμε τις γνωμοδοτήσεις μας, μπορούσαν αυτές να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη, αλλά βεβαίως όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν τρόπον τεινά στο εθνικό επίπεδο, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα μπορεί να διαφέρει. Είναι λοιπόν προφανές για μένα πως ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο έχει προσθέμενη αξία, έχει συστήσει διάφορα δίκτυα και δίνει σαφή στοιχεία. Απ' την άλλη θα ήθελα να σας προσκαλέσω να δούμε μαζί πώς θα μπορούσα να σας πείσω. Τι θα χρειαστεί δηλαδή για εσάς ώστε στο μέλλον να πιστεί η Επιτροπή σας. Γιατί δίνετε πάρα πολλά χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο και θα ήθελα εγώ να χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα χρήματα. Σας προσκαλώ λοιπόν να έρθετε στη Στοκχόλμη αλλά και να συζητήσουμε εδώ πέρα μαζί το πώς ε, θα μπορούσα να σας ε, πίσω στην ε, κίνη αυτή η περίοδο μας. Α, δύσκολη η δουλειά σας, λέει ο Πρόεδρος, σας το υπόσχομαι, αλλά οπωσδήποτε θα αξίσει. Λοιπόν, Άννα Ασπαχ, έχει τον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω κάποια, κάποιες πρακτικές, ε, ρεαλιστικές ε, πρωτοβουλίες κοντά στον πολίτη σε τρεις τομείς που δεν αναφέρατε. Για, την, ε, για τα βακτήρια της φυματίωσης που έχουν απτύξει αντοχή στα αντιβιωτικά γιατί όλο και περισσότερα τέτοια κρούσματα έχουμε από μετανάστες ή από ανθρώπους που ταξιδεύουν στη Ρωσία και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Επίσης, αναφέρατε το επόμενο ζήτημα, αλλά όχι σε μεγάλο βάθος, οι εμβολιασμοί των παιδιών. Όλο και περισσότεροι οι γονείς ε, αποφασίζουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη όταν μιλάμε για τους ε, παραδοσιακού εμβολιασμού όπως το εμβόλιο για την πολιομιελίτιδα, αλλά το ίδιο ισχύει και παροτίτιδα και την ε, ερυθρά. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους γονείς ότι είναι σημαντικό να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο αναφέρατε είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν ρεαλιστικά σχέδια για αυτά τα οποία λέγαμε τροπικές ε, ασθένειες που πλησιάζουν ε, σιγά σιγά π.χ. βλέπουμε ελονοσία και άλλες ασθένειες ε, δάγκιος πυρετός βλέπουμε να ανεβαίνουν πιο βόρεια μπορούμε να κάνουμε κάτι ρεαλιστικά να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και τους γιατρούς για αυτές τις απειλές Thank you very uh, Ευχαριστώ πολύ. Η φυματίωση είναι πράγματι πολύ σημαντική. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στα οποία δίνεται εντύπωση ότι έχουμε ε, φυματίωση, αλλά τα προβλήματα δημιουργούνται στις ευάλωτες ομάδες η αντοχή στα ε, φάρμακα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά τα πάντα ξεκινούν με τη διάγνωση μιας ασθένειας. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη προσφέρει υποστήριξη προκειμένου να γίνεται η σωστή διάγνωση στο, σε σύντομο χρονικό διάστημα και να επιτρέπεται στα εργαστήρια να γίνεται και μια σχετική δοκιμή για την αντοχή σε ε, φάρμακα, σε μικρόβια. Μόνο ένα κλάσμα των ανθρώπων που έχουν αντοχή στα φάρμακα ε, τη χάνουν σωστή διαγνωση και φυσικά χωρίς τη σωστή διάγνωση δεν μπορεί να λάβουν και τη σωστή θεραπεία. Ε, το κέντρο θέλει λοιπόν να προωθήσει τη σωστή κατάρτιση των εργαστηρίων και ελπίζω να μπορέσουμε να λάβουμε και χρηματοδότηση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση των ε, ε, εργαστηρίων, διότι ξέρουμε ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, υπάρχουν πολύ περισσότερα περιστατικά. Δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι ε, λογικό να γίνονται δοκιμές έλεγχη συγγνώμη, σε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν ή σε μετανάστευση. Θέλουμε να είναι σε ε, προτεραιότητα στις εθνικές ε, ατζέντες, ε, φαίνεται ότι ο κόσμος είναι λίγο αδιάφορος όσον αφορά στη φυματίωση και δεν δίνει τη δέουσα προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό να λυθεί η δέουσα ε, προσοχή και να προσέξουμε και τα ε, συστήματα υγείας γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλές ανισότητες στα συστήματα της υγείας υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν πολύ ισχυρό σύστημα υγείας και εκεί υπάρχουν πολλά περιστατικά φυματίωσης και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την ε, φυματίωση. Τώρα για τον εμβολιασμό των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε τους γονείς ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ο εμβολιασμό των παιδιών τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επιδημία ηλαρά στην Ευρώπη. Η ηλαρά στην Ευρώπη είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι η ηλαρά μπορεί να προκαλέσει και θάνατο, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές ε, ασθένειες ως ε, παρενέργεια, όπως η εγκεφαλίτιδα και η πνευμονία. Ξέρουμε ότι η, Ιρλανδ... η... η Λαρά στη Λατινική Αμερική ε, έχει εξαλειφθεί, ενώ στην Ευρώπη δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ενθαρρύνουμε την ανατολική πλευρά της Ευρώπης να κάνει εμβολιασμούς, κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη έχει ένα πολύ καλό σχέδιο στην ιστοσελίδα του. Λέγεται πρόγραμμα Venus ε, είναι ουσιαστικά ένα, ε, μια σελίδα στην οποία μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις πολιτικές ε, υγείας και σας παρακινώ να το δείτε διότι είναι προφανές ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική πολιτική για τον εμβολιασμό των παιδιών. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το πρόγραμμα Βάσκο. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συλλέγονται όλες οι πληροφορίες ε, για τις επικίνδυνες παρενέργειες ε, που σχετίζονται με τον παιδικό εμβολιασμό. Και είναι προφανές ότι ο εμβολιασμός των παιδιών είναι πάρα πολύ ασφαλής και θα πρέπει να πείσουμε τους γονείς ε, δίνοντάς τους τις κατάλληλες ε, πληροφορίες για να εμβυλιάζουν τα παιδιά τους. Και ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να πείσουμε τους γονείς. Ε, ευχαριστώ κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσει μου ακολουθούν μετά την, τις ερωτήσεις της κυρίας Ροτ Μπέρεντ και της κυρίας Γκροστέτ. Όσον αφορά τον εμβολιασμό για τη γρήπη H1N1, περάσαμε μια αρκετά δύσκολη περίοδο και με τη διαχείριση της κρίσης αυτής νομίζω ότι αυξήσαμε την ε, καχυποψία της κοινή γνώμης έναντι των όσων δηλώνονται δημοσίως, έναντι των επιστημονικών οργανισμών και ακόμη και έναντι των αποφάσεων που αναγκαστήκαμε να λάβουμε και ε, για αυτό αυτού του λόγου πολλοί στο Κοινοβούλιο ζητούν μια εξεταστική επιτροπή ακριβώ για αυτό το θέμα. Τέλο πάντων, αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Η ερώτησή μου είναι απλή, κύριε Διευθυντά. Ε, σκοπεύετε να κάνετε σημαντικές τροποποιήσεις όχι μόνο στα θέματα δήλωσης συγκρουόμενων συμφερόντων, αλλά και στη διαχείριση αυτών των συγκρουόμενων συμφερόντων. Δηλαδή, όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να απαγορεύεται σε κάποιον να συμμετάσχει σε κάποια λήψη αποφάσεων και γενικότερα στη διαδικασία που ακολουθείτε διότι σε αρκετούς από εμά ε, φαίνεται ότι η ύψιστη προτεραιότητα είναι να υπάρχει διαφάνεια για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών μας στους κοινοτικούς οργανισμούς, ούτως ώστε στην επόμενη επιδημία να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση, διαφορετικά δεν θα μας πιστεύει κανένας. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για την απάντηση. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ δύσκολο διότι οι εμπειρογνώμονες δραστηριοποιούνται σε πολλά δίκτυα. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι χρειαζόμαστε τις φαρμακοβιομηχανίες, διότι αν δεν υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες δεν θα υπάρχουν και εμβόλια. Όμως, χρειαζόμαστε και μια σαφή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, είτε πληρώνεται κάποιο από μια φαρμακευτική εταιρεία είτε όχι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και δεύτερον, ο πρόεδρο τη Επιτροπή θα πρέπει να κρίνει αν η σύγκρουση συμφερόντων στη δεδομένη περίπτωση είναι αποδεκτή ή όχι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ε, διστάζω ως προς την ε, ε, ξεκάθαρη απόφαση που θα λαμβάνετε επ' αυτού. Νομίζω ότι πρέπει ε, να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση, να είναι ανοιχτά τα πρακτικά, δεν κρύβουμε ούτε τα πρακτικά ούτε τη σύνθεση των επιτροπών και είναι ενδιαφέρον να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από τις αξιολογήσεις, από τις έρευνες που γίνονται τώρα στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη και ίσως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Ζέβε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις ε, που σας απευθύνθηκαν αφορούν κυρίως την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη για την πολιτική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και όταν κάποιος φορέας θέλει να έχει αξιοπιστία ε, θα πρέπει να έχει αξιοπιστία και έναντι των πολιτών και έναντι των εθνικών αρχών. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό το θέμα της εμπιστοσύνη και η κυρία Ροτμπέρεντ και η κυρία Λεπάζ ε, ε, ε, εκφράστηκαν από αυτού του θέματος. Πώς θα εκφράσετε αυτή την αξιοπιστία του οργανισμού τον οποίο προσωπείτε, την αξιοπιστία τη δική σας προσωπικά. Τι δράσεις σκοπεύετε να αναλάβετε. Και ε, δεύτερον, όσον αφορά την γρήπη H1N1, ε, είδαμε σε πολλά κράτη-μέλη ότι χρειάζεται ίσως ένας ευρωπαϊκός συντονισμός για μέτρα πρόληψης. Οι αντιδράσεις στα κράτη-μέλη ήταν ε, κατά πολύ διαφορετικές όσον αφορά την προμήθεια φαρμάκων. Στην Γερμανία παραγγέλθηκαν 40 εκατομμύρια δόσεις, ενώ άλλα κράτη-μέλη επέλεξαν διαφορετική πορεία και ίσως ε, να είχαμε τελικά το ίδιο αποτέλεσμα για, με πολύ μικρότερο κόστος για την προμήθεια φαρμάκων. Μας ενδιαφέρει ε, με, την ισχύουσα, με τις ισχύουσες αρμοδιότητες ε, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους πολίτες μας. Και ένα θέμα που ανέφερε και ο συνάδελφος Λίζε αφορά το νερό και πάλι. ιδίως ε, για ε, νόσους που μεταδίδονται μέσα από το νερό, νομίζω ότι ίσως να χρειάζεται κάποια βάση δεδομένων. Υπάρχουν ε, στατιστικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν και για τις μελλοντικές, να λαμβάνουμε υπόψη και τις μελλοντικές αλλαγές του κλίματος, ούτως ώστε να έχουμε την λήψη των κατάλληλων μέτρων. Ευχαριστώ πολύ και ο κ. Ζέμπερ ενδιαφέρεται για το νερό. Απάντηση. Λέτε ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των διαφόρων οργανισμών. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να υπερασπίσω το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης με αυτά που λέω. Βλέποντας την τωρινή κατάσταση, Και διαβάζοντας και πάλι την ομιλία που έκανε ε, η Διευθύντρια εδώ το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι η πρόβλεψη ήταν πολύ ισορροπημένη. Δεν ανήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης δραματικά σενάρια. Η Σουζάννα ε, Γιάκομ πολύ σαφώς έκανε την αξιολόγησή της. Καθώς εγώ βλέπω, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης δίνει και σε εσά και στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές. Από αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία. Και στο μέλλον θα ήθελα να επαυξήσω ακριβώς αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Έχουμε πολύ καλούς εμπειρογνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφέρω τα ονόματα. Είναι εξαιρετικοί χωρίς να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, διστάζω κάπως και σε κάτι ακόμη. Και βέβαια είδα το τι συνέβη στα διάφορα κράτη-μέλη. Και κάπως εξεπλάγην από τις διαφορετικές αντιδράσεις. Όμως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του κινδύνου. Βεβαίως έχει ένα ρόλο το Συμβούλιο και μπορώ να σας δώσω τη δική μου προσωπικά και μόνο γνώμη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσει πολλά χρήματα εάν τα κράτη-μέλη ήταν πρόθυμα να έχουν περισσότερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Αλλά αυτό δεν είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης, είναι ρόλος των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να δίνουμε τις επιστημονικές ε, αποδείξεις ότι είναι ασφαλές να γίνει το εμβολιασμός, ότι είναι ασφαλές για κάποιες ομάδες ηλικιών κλπ. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το νερό, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε στοιχεία και αυτό έχει σχέση και με άλλη ερώτηση. Χρειαζόμαστε εμπειρογνωμοσύνη για να κάνουμε τη διάγνωση των λοιμόξεων που μεταδίδονται μέσα από το νερό. Δεν είμαστε ακόμη επαρκώ εξοπλισμένοι γι' αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη έχει πολλέ πρωτοβουλίε, ούτω ώστε να επιμορφώσει τα εργαστήρια και να κάνουν τη σωστή διάγνωση και για το νερό. Και θα είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες λοιμώξεις από το νερό ή από τα τρόφιμα ή άλλους, άλλες περιβαλλοντικές πηγές. Άρα είναι ένα θέμα που παραμένει στην ημερήσια διάταξή μας. Και τώρα, ο κύριος Κυλακάκης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κλεγμένη Πρόεδρε, έχω Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη ήδη αναφέρθηκε και αφορά την ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Το θεωρείτε κίνδυνο. Πώς παρακολουθείτε την αύξηση της ε, αντίστασης αυτής και ειδικά εκεί όπου είναι πιο προφανές. Γιατί στην περίπτωση αυτή βεβαίως η άμυνά μας ε, είναι τόσο καλή όσο το χειρότερο σημείο και όχι το καλύτερο σημείο. Και πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε, γιατί κάποια στιγμή θα μπορούσε να είναι ε, θανάσιμος κίνδυνος ε, για τον πληθυσμό της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό σύστημα. Το δεύτερο ερώτημά μου προέρχεται από το ότι είμαι οικονομολόγος. Θεωρείτε πως τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας συνολικά επενδύουν ε, βέλτιστα από οικονομική σκοπιά όσον αφορά την πρόληψη λιμωδών ασθενειών και αν όχι πώς σκοπεύετε ε, να, να βοηθήσετε στη βελτίωση της ε, πρόληψης ε, ως μία επένδυση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Υγείας και της Ευρωπαϊκής Οικονομίας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η... Αντίστοιχα, αντιμικροβιακά πράγματι είναι κίνδυνος, πρέπει να επιτηρήσουμε σε διαφορετικά πεδία πρώτα απ' όλα στα νοσοκομεία. Υπάρχει λοιπόν το δίκτυο Earsnet, το οποίο αφορά ακριβώς την ε, αντίσταση στα αντιμικροβιακά αντιβιωτικά, αλλά βεβαίως ε, ίσως πιο σημαντικός είναι ο τομέας της κτηνιατρικής, της γεωργίας. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερα σε αυτόν τον τομέα και στην παρακολούθηση της αντίστασης ε, τον Και χαίρομαι για την πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν που λέγεται «Ένας κόσμος, μία υγεία» και συνδυάζει την ιατρική με την κτηνιατρική. Και τώρα χρησιμοποιούνται πολλά κτηνιατρικά αντιβιωτικά και πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέπειε έχει αυτό. Ο τρίτος πυλώνας είναι η χρήση των αντιβιωτικών. Γνωρίζουμε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης αντιβιωτικών και της αντίστασης, όσο περισσότερο η χρήση τόσο μεγαλύτερη αντίσταση και αυτές οι τρεις ε, πηγές ε, πληροφόρησης ε, πρέπει νομίζω να κατευθύνουν την πολιτική μας. Γνωρίζω πως το κέντρο δίνει αυτές τις κατευθύνσεις, γνωρίζω επειδή εγώ είμαι μικροβιολόγος, πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε συγκρίσιμα δεδομένα, οπότε πρέπει να επενδύσουμε και στην εργαστηριακή πλευρά μέτρησης της αντίστασης αυτής, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για το το κάνει αυτό το κέντρο μας και χαρικά επίσης για το ότι ήταν υψηλή προτεραιότητα αυτό το θέμα. Νομίζω πως πέρσι είχατε μια εκδήλωση για την σωστή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Οπότε γνωρίζετε το πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τις ε, επενδύσεις ε, στην υγεία, πριν από ένα μήνα υπό την ιδιότητά μου ως ε, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου πρότεινα να επενδύσουμε περισσότερα στην ε, δημοσιογεία, όχι μόνο στις λοιμώδεις ασθένειες νόσους, αλλά και στην παχυσαρκία, τη σωματική δραστηριότητα κτλ. Αξίζει, μπορώ να σας το αποδείξω, ε, να επενδύσουμε στις λοιμώδεις νόσους, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδύσουμε ξανά στην ε, φυματίωση, στον εμβολιασμό των παιδιών, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ήταν πρόφανες και από την επιδημία της γρήπης πως ε, ε, είχε πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες. Και είναι σημαντικό να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες, σχέδια ανάγκης και ελπίζω πως οι πολιτικοί θα πιστούν να επενδύσουν στη δημοσία υγεία και Χόρστ Σνέλχα τελευταίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπρέγγε, έχω κάποιες ερωτήσεις για αυτό το οποίο... Ε, θα ήθελα όμως να επανέλθω σε αυτό το οποίο μόλις είπατε, ειδικά στον αφορά την αντίσταση στα αντιβιωτικά και είπατε πως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την ε, κτηνιατρική πριν από λίγα χρόνια εμείς ρυθμίσαμε τη χρήση αντιβιωτικών ε, στα ζώα έτσι ώστε να είναι διαφορετική η δομή και η χρήση. Οπότε μην ξεχνάτε πως ε, ειδικά στα νοσοκομεία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης της αντίστασης. Και στο πλαίσιο αυτό δύο πράγματα ακόμα, γιατί αναφέρατε την κλιματική αλλαγή και γνωρίζετε πως αυξάνεται τα ταξίδια και με τις ασθένειες που εμφανίζονται στις περιοχές μας ε, κατά 57% από όσο γνωρίζω μιλάμε για για ζωονόσους που βεβαίως πλήττουν και το ζωικό κεφάλαιο αλλά μεταφέρονται και σε ανθρώπους. Οπότε σκοπεύετε να συνεργαστείτε τόσο στενά με την κτηνιατρική έτσι ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε πολύ νωρίτερα αν έρχονται ε, ασθένειες από την Αφρική στον, στον νότο της Ευρώπης και πώς το βλέπετε, δεν το βλέπω καθόλου απλό. Επίσης μιλήσατε για την παχυσαρκία. Το Κοινοβούλιο βεβαίως ε, τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την ε, καταπολέμηση της ε, παχυσαρκίας και δεν ξέρω, εγώ είμαι κάπως απεσιόδοξος ε, για το αν θα τα καταφέρουμε, αλλά ίσως μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα, να μας εξηγήσετε δηλαδή εσείς πώς φαντάζεστε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, να επηρεάσουμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, ειδικά των νέων, έτσι ώστε να δοθεί μια σαφής κατευθυντήρια γραμμή. Ποια θα είναι η στρατηγική υγείας της Κομισιόν. Καθώς ε, ε, επίσης και όσον αφορά αυτή την αλλαγή σε σχέση με τους ε, εμβολιασμούς και τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Χαίρομαι που αναφέρεστε και στη σχέση μεταξύ, κτηνιατρικού και ανθρώπινου κόσμου. Έχω μιλήσει και με τον επικεφαλής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων και πραγματικά θα ήθελα να είναι πιο στενές οι σχέσεις μας και ελπίζω και στο μέλλον να υπάρχουν και ενοποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μια κοινή όπως την αποκαλείτε εσείς επιστημονική άποψη. Αυτό θα ήταν ευτυχές. Ε, θα ήθελα να μάθω περισσότερα, ε, μια και είπατε ότι έχετε ήδη συζητήσει το θέμα της χρήσης ε, αντιβιωτικών ε, στην κτηνιατρική και θα με ενδιαφέρει να μάθω περισσότερα. Όπως σας είπα και πριν, η παχυσερκία δεν είναι στην εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Πρόληψη, αλλά θα μπορούσα να σας πω και λίγα λόγια επί του θέματος. Είναι ιδιαίτερος δύσκολο να γνωρίζει κάποιους πράγματα, να εκπαιδεύει ε, κάποιους για την υγεία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επικοινωνία και στην εντολή του κέντρου για, την, ε, για τον εμβολιασμό ε, των παιδιών και για το νιό των κονδυλωμάτων που αφορά τις γυναίκες. και πραγματικά πιστεύω ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την ε, ε, παιδεία, για την υγεία. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα σχολεία. Ελπίζω, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην εντολή του κέντρου, να προσπαθήσουμε να επενδύσουμε περισσότερο σε, μια πιο, σε ένα πιο υγιή τρόπο ζωής ε, και να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση στα σχολεία, να μπορέσουν να τα συμπεριλάβουν στο σχολικό πρόγραμμα. Και τελευταία ερώτηση, για τρίτη φορά δίνω το λόγο στην Dagmar. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι για την πολλαπλή αντίσταση στα βακτήρια. Ε, ρώτησαν και οι συνάδελφοι σχετικά με την οικονομική επίπτωση. Χρειαζόμαστε πολλές φορές νέα αντιβιωτικά, χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία, που θα αφορά τα αντιβιωτικά. Πρέπει να δώσουμε νέα κίνητρα. Ίσως αυτό να είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου των Φαρμάκων, του EMEA. Μήπως θα μπορούσαμε να διδαχθούμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων ε, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ε, και όσον αφορά τις γλυκαντικές ουσίες θα, θα πρέπει ε, να ξέρουμε ποιοι είναι τα μέλη και οι επικεφαλής αυτών των ομάδων που ασχολούνται με θέματα τέτοια. Ε, θα μπορούσατε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι εταίροι σας ε, στη συνεργασία είναι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, γιατί εσείς δεν είστε εταίρεος των κρατών μελών, είστε εταίρεος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, όχι του Συμβουλίου δηλαδή. Επομένως θα πρέπει να συμβουλεύεστε, θα πρέπει να έχετε να συμβουλεύετε την Επιτροπή, όπως θα θέματα της γρήπης των χείρων παραδείγματος χάρη. θα περάσετε από ένα εθνικό Ινστιτούτο, ένα μεγάλο Ινστιτούτο όπως είπατε, σε ένα οργανισμό που θα πρέπει να δίνει και συστάσεις ε, και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι όντως μπορείτε να εκπληρώσετε αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Κατά την παρουσίασή μου για την εκλογή μου, ανέφερα ότι η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο λόγω περιεχομένου, αλλά και για επιχειρησιακούς σκοπούς. Και μία από τις πτυχές ε, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα θέματα διασφάλισης ποιότητας, γιατί η διασφάλιση ποιότητας είναι και αυτή ένα σημαντικό θέμα και ξέρω ότι όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και τα ίδια διλήμματα. Θα ήθελα λοιπόν να επενδύσουμε στη σχέση με όλους αυτούς τους άλλους οργανισμούς και όχι να επανεφεύρουμε εμείς τον τροχό. Πρώτη φορά εμφανίζομαι εγώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ίσως γνωρίζετε ότι στο εθνικό μας σύστημα ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε άμεσα με το Κοινοβούλιο. Καλέσαμε διάφορα κόμματα του Κοινοβουλίου να επισκεφθούν το Ινστιτούτο μας και μάλιστα ζήτησε και κάποιο κοινοβούλιο, ε, κάποιο κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφθεί το Ινστιτούτο μας και με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε σε αυτό το αίτημα. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας και να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες και πώς θα μπορούσαμε εμείς ως ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης να εξυπηρετήσουμε αυτά τα οποία εσείς θέλετε. Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και από δύο εκπροσώπους του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτοί φέρουν την ευθύνη για το πρόγραμμα εργασιών μας. Θα ήθελα όμως να έχουμε συζητήσεις και σήμερα είναι η αρχή αυτών των συζητήσεων. Θα επιθυμούσα πολλές φορές να επαναλάβω τέτοιες επισκέψεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις. Η πρώτη σας επίσκεψη στο Κοινοβούλιο, όπως ε, είδαμε, ε, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερο δυναμισμό και ήταν πολύ ζωντανή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που επισκεφθήκατε την ε, Επιτροπή μας. Στις 5 έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Θα αξιολογήσουμε και αυτά τα οποία είπαμε. Θα στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και ε, κλείνει η συνεδρίαση. Θα συνεδριάσουν οι συντονιστές στις 5.